για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Bienvenido, señor comisario. Tiene usted la palabra. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη, εκ μέρου του Επιτρόπου του κυρίου Κανιέτε, καταρχάς σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Λευκορωσία. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω σχετικά με το πώς εργαζόμεθα για την εξασφάλιση του ότι θα επικρατούν τα μεγαλύτερα επίπεδα ασφαλείας στις καταστάσεις αυτές. Η πυρηνική ασφάλεια παραμένει η βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επιβεβαιώνει αυτό και η στρατηγική πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση. Θέλουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία, θέλουμε να επικρατεί διαφάνεια, να υπάρχει εμπιστοσύνη και χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε τον ύψιστο δυνατό βαθμό ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο η ασφάλεια. Τώρα τη συνεργασία για την πυρηνική ασφάλεια με τη Λευκορωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση Λευκορωσία. Πάντα ακολουθούσαμε τη συγκεκριμένη προσέγγιση με τη Λευκορωσία πυρηνική ασφάλεια και η προστασία η ιδεολογική ήταν βασικός στόχος των συνομιλιών μας. Από το 2011 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήχε στην Λευκορωσία και στις αρμόδιες αρχές τεχνική αρρωγή σύμφωνα με το μέσο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Πυρηνική Ασφάλεια διαβιβάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στο ρυθμιστικό επίπεδο στη Λευκορωσία το σύστημα αδειοδότησης, τις συνθήκες αδειοδότησης και ελέγχων, επιλογή επίσης τοποθεσιών της εγκαταστάσης και τη λειτουργία αυτών. Από τον Απρίλιο του 2015, ένας εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βρίσκεται στο Μίνσκ. Εκεί ενισχύουμε τον αρμόδιο φορέα για την κατασκευή πυρηνικής εγκατάστασης από το αρχικό στάδιο Απότερο στόχο είναι η τεχνογνωσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να βοηθήσει τη Λευκορωσία. Να μπορεί να συμμορφώνεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρότυπα η Λευκορωσία. Μέσω της τεχνικής βοηθείας, η αρμόδια αριθμιστική αρχή της Λευκορωσίας έχει βελτιώσει το ανθρώπινο και τεχνικό υλικό τη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα της Λευκορωσίας πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και χρειάζεται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων. Τώρα για την πυρηνική ασφάλεια και τις δοκιμές αντοχής. Όπως προανέφερα, χρειάζεται ανοιχτή προσέγγιση και διαφάνεια. Είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την πυρηνική ασφάλεια. Χρειάζεται συνεργασία με τους γειτονές μας. Πρέπει να συνεργαζόμαστε ανοιχτά. Αυτό θα είναι υποφελέ και για τι δύο πλευρέ, λόγω ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσία. Και θα δημιουργείται και κλίμα εμπιστοσύνη. Σε αυτό το πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την εκτεταμένη χρήση πλευρά Δευκορωσία, τη τεχνογνωσία, τη αρμόδια και ε, υπηρεσία για την πυρηνική ανέργεια, ούτω ώστε να εξασφαλίσει τη ασφάλεια. Πριν αναφερθώ στο που βρισκόμαστε όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής στο Στρόβετς να τονίσω δύο πράγματα. Είναι στοιχεία σημαντικά για να κατανοήσουμε την όλη διαδικασία. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι οι δοκιμές αντοχής όσον αφορά τις πυρηνικές εγκατάστασεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες διεξάγονται εθελοντικά. Νομικώς πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να υποχρεώσει κανένα κάτω μέλος ούτε τρίτη χώρα που επιλέγουν την πυρηνική ενέργεια να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους δοκιμές αντοχής. Όμως υπάρχει μια πολιτική δέσμευση για δοκιμές αντοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ενθαρρύνουμε να επεκταθούν αυτές οι δοκιμές και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είχαμε έκκληση του Μαρτίου του 2011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζητάει συνεργασία, διαφάνεια, αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τι πυρηνικέ εγκαταστάσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά ζητεί το Συμβούλιο να γίνονται παρόμοιε δοκιμέ αντοχή και σε γειτονικέ χώρε και παγκοσμίω. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πραγματοποίηση δοκιμών αντοχή σε γειτονικέ χώρε. Είναι ενθαρρυντικό το ότι η Ουκρανία ήδη εθελοντικός έχει συμμετάσχει σε τέτοια εγχειρήματα και η Αρμενία ακολουθεί τώρα τη διαδικασία να το πραγματοποιήσει αυτό με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, οι δοκιμές αντοχής είναι εθνική αρμοδιότητα. Διεξάγεται από τον αρμόδιο φορέα και την αρμόδια εποπτική ρυθμιστική αρχή της χώρας. Μόνο αφού γίνουν οι εξολογήσεις από δοκιμές αντοχής σε εθνικό επίπεδο, γίνεται εξολόγηση και ενημερώνεται δεόντως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάνει εξακριβώσεις και παληθεύσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επαφή με τι αρμόδιε εθνικές αρχές. Τον Ιούνιο του 2011, βάσει Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκετές χώρε, χώρες, τη Λευκορωσία, εξέφρασαν την επιθυμία τους να πραγματοποιήσουν δοκιμές αντοχής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις υπογράφοντας μια δήλωση για την διεξαγωγή αυτών των δοκιμών αντοχής. Έκτοτε, παροτρύνουμε τη Λευκορωσία να πραγματοποιεί τέτοιες ε, δοκιμές αντοχής των πυρηνικών εγκαταστάσεων υπηρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το φως των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2016 ότι η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ενώσεως Λευκορωσίας θα εξελιχθεί θετικώς και σε αυτό το τομέα δηλαδή των δοκιμών αντοχής. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Λευκορωσία ότι τώρα έχει δημιουργήσει ένα νομικό μέσο που διευθετεί την εφαρμογή αυτών των δοκιμών αντοχή στι πυρηνικέ εγκαταστάσει και ευθυγραμμίζεται με τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Η Λευκορωσία επίση ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών στο Στρόβετς θα ετοιμαστεί έκθεση αξιολόγηση. Θα υποβληθεί αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την διάρκεια του 2016 και του 2017 από την πλευρά μας. Κάνουμε αναγκαίες προετοιμασίες για τον έλεγχο ομοτήμων έχουν γίνει προετοιμασίες. Και τώρα συμπεριλαμβάνεται αυτό στο πρόγραμμα εργασίας των ρυθμιστικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η ομάδα των εμπειρογνωμόνων των Ευρωπαίων θα διοργανώσει τον, τον έλεγχο μοτίμων από τη στιγμή που θα παραλάβουμε την έκθεση της Εθνικής Αξιολογήσεως. Αυτό είναι θετικό βήμα μεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες οι αναγκαίες στην Λευκορωσία ε, και να εξασφαλίζεται ότι θα υποβληθεί η έκθεση για τις δοκιμές αντοχής στο ταχύτερο δυνατόν. Γι' αυτό οι υπηρεσίες μας σχεδιάζουν τεχνική αποστολή στη Λευκορωσία τους επόμενους μήνες, ούτω ώστε να συζητήσουν την επιτευχθήσα πρόοδο. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην αύξηση της ευαισθησίας της Λευκορωσίας αφορά την πυρηνική ασφάλεια και να το συζητά αυτό σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Θα συνεχίζουμε να προωθούμε το ύψιστο επίπεδο προδιαγραφών όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια στη Λευκορωσία μαζί με όλους τους διεθνείς μας εταίρους. Επιτρέψτε μου επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε στενές επαφές με τα γειτονικά κράτη-μέλη, κυρίως με τη Λιθουανία, για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό, το Στρόβε. Σας διαβεβαιώνω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως όσον αφορά τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Στυλιανίδη. Αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Μάμκινς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πυρηνικό σταθμό τη ε, Λευκορωσία είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται το 1980 όμω. Λόγω του Τσερνομπίλ το 1986 τα σχέδια καθυστέρησαν και υλοποιήθηκαν πριν από μία δεκαετία μόλις. Είχε ξεκινήσει η κατασκευή του 2013 και αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αντιδραστήρας αυτός, ε, ύδατος, ε, είναι ο ίδιος ο οποίος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και στο Χαρχικίδη στην Φιλανδία. Οι φόβοι της διεθνούς κοινότητας, ειδικά της Λιθουανίας, είναι κατανοητή. Η Λευκορωσία δεν είχε ποτέ πυρηνική ενέργεια στο εδαφός της και άρα τίθεται ζήτημα αδυναμίας να λειτουργήσει σωστά το εργοστάσιο. Οπότε για να ανακουφιστούν αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει η Λευκορωσία να επιτρέψει κάποια, κάποιες δοκιμές υπό την αιγίδα της ε, Διεθνούς υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας καθώς επίσης και μια αξιολόγηση περιβαλλοντικών αντικτύπων, ειδικά όσον αφορά τα πόσιμα νερά και τις πηγές που εκβάλλουν στην Λιθουανία. Βεβαίω τώρα που έχουν αρθεί οι κυρώσεις, οι σχέσεις μας αναθερμαίνονται, οπότε νομίζω πως μια λύση για το πυρηνικό εργοστάσιο του Όστροβετ θα βρεθεί σύντομα, καθώς δεν μπορεί παρά να υπάρξει μια λύση η οποία θα είναι μια λύση πολυμερούς συνεργασίας με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα. Λευκορωσία, Λιθουανία, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε άλλο διεθνές θεσμικό όργανο. Και θα ήθελα να προσθέσω πως η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον με την σωστή συντήρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φωτίγα. Σας ευχαριστώ. E, Μιλάμε ε, ε, για το ε, Τσερνομπίλ, για την αρχή του τέλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 23% του επίπεδου πεδάφους της Λευκορωσίας έχει μολυνθεί. Επειδή πρόκειται όμως για πυρηνική ενέργεια, κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθεί μία συντηρητική πολιτική. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις πυρηνικές μονάδες. Στη συνέχεια όμως η Λευκορωσία άλλαξε πολιτική και τώρα θέλει να συμμετάσχει στα γενικότερα πλαίσια στη γενικότερη πολιτική της περιοχής. Το Όστροβιέτς αποτελούσε μία κοινή προσπάθεια της Λευκορωσίας με τη Ρωσία με, ένα μικρό, με μία μικρή συμμετοχή της Φιλανδίας. Το Όστροβιτς βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας πολύ κοντά στα σύνορα Λιθουανίας και Λευκορωσίας και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και κίνδυνος σεισμικών δονήσεων. Υπάρχει και ε, ένας ε, εναέριος διάδρομος. Αυτός ο διάδρομος ε, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει. Αυτός ο αεροδιάδρομος που περνάει πάνω από το εργοστάσιο αυτό. Θεωρούμε ότι η Λευκορωσία δεν τήρησε τη, όλες τις υποχρεώσεις των διεθνών συμβάσεων και δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό τον φύλακο μένουν και Πολωνοί οι οποίοι είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Θα μιλήσω λιθουανικά, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Εδώ και αρκετά μερικά χρόνια είχε δηλωθεί ότι ο πυρηνικός σταθμός του Όστροβιτς θα πρέπει να είναι ο φθηνότερος που έχει κατασκευαστεί από τους Ρώσους οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό είχε παρατεθεί σε μια ομιλία ηγέτου. Ακούγοντάς το αυτό, τρομάζω και ανατριχιάζω και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι ήρεμος. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν αληθές. Ο πυρηνικός σταθμός του Όστροβετς κατασκευάζεται με έναν τρόπο θα έλεγα καταφριστικό και γίνεται, γίνονται οικονομίες εις βάρος της ασφαλείας. Οι διεθνείς ασφα... ε, συνθήκες ασφαλείας παραβιάζονται. Δεν γίνονται οι αναγκαίες δοκιμές αντοχής και γίνονται και ε, κάποιες κλοπές όσον αφορά το υλικό. Κατασκευάστε στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση 50, 50 χιλιόμετρα από το Βίλνιους. Είναι κάτι παράνομο και ανασφαλές σαν κατασκευή. Σήμερα ακούμε κάποιε εξηγήσει που μα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά λυπάμαι, κύριε Επίτροπε, αυτά που μα είπατε δεν αρκούν. Η απόφαση να κατασκευαστεί ο πυρηνικό σταθμό Σταστοβίτ ήταν πολιτική απόφαση τη Μόσχας η απόφαση να παραμείνει η παραγωγή ενέργεια στην περιοχή. Πρέπει να ξυπνήσουμε πριν είναι πολύ αργά. Ο συμβιβασμό όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια είναι κάτι που οδηγεί στην καταστροφή. Αντιμετωπίζουμε τον δικτάτορα Λουκασέγκο που προσπαθεί να κατασκευάσει ένα πυρηνικό κράτο. Δεν έμαθε τα μαθήματα του Τσερνόμπιλ. Κυρίε και κύριοι, μάθαμε εμεί τα μαθήματα του Τσερνόμπιλ. Θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλου ότι οι πυρηνικέ καταστροφέ δεν γνωρίζουν σύνορα. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μία λύση εφικτή. Αυτή η παράνομη κατασκευή πρέπει να σταματήσει. Το πρόγραμμα Ωστροβίτς θα μπορούσε να ε, προωθηθεί μόνο αν υπήρχε ο κατάλληλο διάλογο που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει και του σύνεγγυ στη αυστηρότητα την κατασκευή. Χρειαζόμαστε μια καλή αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ενώση που απευθύνεται προ το Μίνσκ και τη Μόσχα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη την επιρροή μα. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία ε, των συνομιλιών με το Ιράν όταν μιλάμε τη Λευκορωσία. Συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΙΕ. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι γιατί μπορώ να λάβω το λόγο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η ασφάλεια των πυρηνικών μονάδων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται στα σύνορα, στα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 440 νέοι αντιδραστήρες έχουν αρχίσει να λειτουργούν και θα δημιουργηθούν και άλλοι 133 και σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, στα πλαίσια της επαιτίου για το Τσερνομπίλ ζήτησα να γίνει μία ημερίδα με εμπειρογνώμονες για να αντιλήσουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η μονάδα αυτή πληρεί τους διεθνείς όρους και εποπτεύεται και από ΜΚΟ. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μας απασχολήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα παλαιά κράτη-μέλη μέσα εισαγωγικά, όπως το Βέλγιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προλάβουμε τους κινδύνους. Ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να λάβετε μέρος σε αυτή την συζήτηση. Δυστυχώς απογοητεύτηκα από το ότι ε, Επίτροπος Καλνιέτε δεν βρήκε την ευκαιρία να έρθει να απαντήσει εδώ πέρα σε θέματα αρμοδιότητός του. Για θέματα δηλαδή κινδύνο από τα πυρηνικά εργοστάσια πάρα πολύ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον απογοητεύομαι από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή του εργοστασίου στο Όστροβετς που γίνεται κατά παράβαση διαφόρων διεθνών προδιαγραφών. Τα μηνύματα της Κομισιόν είναι τελείως τυπικά. Πρώτα απ' όλα υπήρχε η προηγούμενη απάντηση του κυρίου Κανιέτε ότι έχουν γίνει δηλαδή ε, τεστ στο νέο πυρηνικό εργοστάσιο παρά το ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και βεβαίως ε, βλέπουμε και την απάντηση του κυρίου Έντρου πώς η Λευκορωσία συμ... συμμορφώνεται με όλες τις διεθνείς ε, συμβάσεις. Εννοώ η σύμβαση του Άρχους και άλλες παραβιάζονται ξεκάθαρα. Η Λευκορωσία αγνοεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Αλλά η Κομισιόν γιατί κάνει τα στραβά μάτια. Ποιος, η οποία Κομισιόν είναι μέλος αυτών των ε, συμβάσεων. Πρέπει να αντιληφθείτε τις ανησυχίες μας. Χτίζεται πυρηνικό εργοστάσιο στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λιθουανίας από ένα αυταρχικό καθεστώς με δάκτυλο Ρωσίας και δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές επιπλέον. Γνωρίζουμε τι, πώς εργάζονται και τι αντίληψη έχουν για τη διαφάνεια. Τον Απρίλιο παραδείγματο χάρη υπήρχε ατύχημα, έπεσε μέρος ε, του κτηρίου αλλά το Μίνσκ το απέκρυψε. Και βεβαίως ε, και το σημείο του εργοταξίου ε, επελέγει πρόχειρα. Δεν προσκάλεσαν τους ειδικού της Υπηρεσίας Ατομικής ε, Ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία αδιαφάνειας. Η Λευκορωσία δεν έκανε αξιολόγηση αντικτύπου για τους ποταμούς που εκβάλλουν στη Λιθουανία ή ένα τεστ αντοχής σε πρόσκουση αεροπλάνου ή ούτε καν σεισμολογικά στοιχεία. Και μόλις τώρα η Κομισιόν αναγνώρισε πως η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της χώρας δεν είναι ανεξάρτητη. Άρα η πυρηνική ασφάλεια δεν εξαρτάται από τους ειδικού, αλλά από την κυβέρνηση μιας αντιδημοκρατικής κιόλα χώρας. Οπότε θα ήθελα η Κομισιόν να καταθέσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να συμμορφωθεί η Λευκορωσία με όλες ε, τις ε, διεθνείς προδιαγραφές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο μήνυμα στο Μίνσκ ότι δηλαδή το περνικό αυτό εργοστάσιο που χτίστηκε χωρίς μέτρα ασφαλείας παραβιάζει όλες τις σχετικές αρχές και δεν επιθυμούμε και ενέργεια από αυτό το εργοστάσιο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ροπέ, έχετε μια μπλε κάρτα με τον κύριο Άρνοτ. Την δέχεστε? Ναι. Κύριε Άρνοτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται βεβαίω για ένα ζήτημα το οποίο είναι ευρύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διεθνές. Είπατε πολλά πράγματα για το τι θέλετε να κάνει η Κομισιόν. Επίσης, αναφέρατε την, τον Διεθνή Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας. Δεν κάνετε όμως κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Τι θέλετε να κάνει ο Διεθνής Οργανισμός Ποινική Ενέργειας. Μπορείτε να μας κάνετε καμία πρόταση. Τι παραπάνω μπορούν να κάνουν δηλαδή. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Πρώτα απ' όλα. Η περιοχή επελέγει, αλλά μετά μόνο σκέφτηκαν να καλέσουν τους ειδικού να δουν αν είναι κατάλληλο το σημείο. Είναι πολιτικές δηλαδή αποφάσεις. Το γεγονός ότι η Λευκορωσία υπόσχεται να κάνει τεστ αντοχής αλλά δεν το κάνει. Και το ότι παραπλανούν την Κομισιόν συνεχώς. Ο Επίτροπος είπε παραδείγματο χάρη πως έχουν ήδη γίνει στρες τεστ. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις ε, λοιπόν που πρέπει να γίνουν σεβαστές γιατί μετά θα υποφέρουμε, θα, αλλά θα έχει γίνει η καταστροφή. Κύριε Έστριτζ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Η Διεθνή Οργάνωση Πυρηνική Ενέργεια παρακολουθεί σε όλο τον κόσμο τεκτενόμενα την πυρηνική ενέργεια από την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτή είναι σαφή περίπτωση όπου η, θα, ότι θα παίξει το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αναπτύξει την ε, πυρηνική ενέργεια, η Λευκορωσία προβληματίσει του γείτονε, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντεθεί στη Διεθνή Οργάνωση για την Πυρηνική Ενέργεια και στον ΟΗΕ. Προφανώ η Λευκορωσία και οδήποτε άλλη χώρα που επιθυμεί να αναπτύξει πυρηνικό τομέα θα πρέπει να υπόκειται σε διεθνεί κανόνες που ισχύουν. Εγώ προσωπικό περισσότερη πυρηνική ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιμένω οι δικέ μα εξελίξει να υπόκεινται ε, στου κανόνε τη Διεθνή Οργανώση Πυρηνική Ενεργεία όπω και κάθε άλλη χώρα. Κυρίαρχα κράτη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αναπτύξουν τις χώρες όσο επιθυμούν από, το, από τη στιγμή που συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες. Αν παραβιάζεται ο διεθνής νόμος, αυτό είναι κάτι που αφορά τον ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επηρεάσει, θέλει να έχει εξουσία. Η εμπορική και η οικονομική συνεργασία είναι μια δικαιολογία για την ύπαρξη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι λόγο για την ύπαρξη. Δεν αρκείται στο να παρεμβαίνει στη ζωή των πολιτών και αυτό ο φορέα απελπισμένα θέλει να παρέμβει στι πολιτικέ των γειτονικών χωρών. Καθένα από εσά, σαν κράτη εθνικά κράτη πρέπει να υποστηρίζετε το Διεθνή Οργάνωση Πυρηνική Ενεργεία και να αντισταθείτε στον πειρασμό να παρεμβαίνετε και να ανακατευόσαστε στα θέματα κυριάρχων ανεξαρτήτων κρατών. Να χρησιμοποιήσετε το, το διεθνέ δίκαιο και αν παραβιάζετε το Διεθνές δίκαιο, αν παραβιάζετε, χρησιμοποιήστε τον ΟΗΕ. Αυτές είναι οι συμβάσει που πρέπει να σέβονται όλα τα κυρίαρχα κράτη και να τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει καμία απέτηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω να κάνει αυτό που κάνει και να δράσει σαν ένα ενίο φορέα, σαν ιονή υπερδύναμη ομοσπονδιακό κράτο. Δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κατάλληλοι φορεί να επιβάλλουν του νόμου αν παραβιάζονται σε τόσο σημαντικό ζήτημα όπω είναι η πυρηνική ενέργεια ε, τότε ας χρησιμοποιήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη, ας χρησιμοποιήσουμε τις εφιστάμενες αρχές και να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται οι λαοί σωστά όσο ενδείκνεται χωρίς να επηρεάζουμε οι πολιτικές φιλοδοξίες και οι πολιτικοί ελιγμοί να παρεμβαίνουν καθιονδήποτε τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κ. Λεμπρετούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πυρηνικές καταστροφές είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές κατά της ανθρωπότητας. Η... Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 και της Φουκουσίμα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει η ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό του Όστροβέτς που ε, θα έπρεπε να τεθεί σε λειτουργία το 2018. Από όσο γνωρίζουμε δεν μπορεί να... Ε, δεν πληρεί μάλλον τα κριτήρια των ε, πυρηνικών αντοχών των δοκιμασιών αυτών και αυτό το βλέπουμε σε 20 αντιδραστήρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα πλαίσιο ασφάλειας που υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα έπρεπε να τηρεί και η Λευκορωσία. Το Όστροβετς βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από το Βίλνιους την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα, τα δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού πυρηνικής ενέργειας. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί μέσα στα πλαίσια της μιμίας μάλλον Ευρώπης των Εθνών. Η ασφάλεια στο Όστροβετς όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Λευκορωσίας. Μην ξεχνάμε ότι το 2015 υπήρχε ένα στρατιωτικό σταθμός ο οποίος λειτουργήσε και βοήθησε και η Ρωσία για την κατασκευή του Όστροβετς. Μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να επιδεινώσουμε τις σχέσεις μας περαιτέρω με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ε, διάφοροι τύποι αντιδραστήρων, ε, πιο δαπανηροί ή λιγότερο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά ατυχήματα θα πρέπει να ε, δούμε κατά πόσο ε, υπάρχουν αντιδραστήρες που πληρούν όλες τις ε, συνθήκες τη στιγμή που λέμε ότι στο Όστρεβιτς δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Στην ουσία εφόσον καταφερόμαστε κατά του Λουκασένκο εδώ και χρόνια, τι κάνουμε. Τον ρίχνουμε στην αγκαλιά της Ρωσίας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Η Ρωσία είναι ο μοναδικός της σύμμαχος και εμείς εξωθούμε αυτή τη ε, συμμαχία. Ο κύριος Ζωρίνιο. Κύριε Επίτροπε, Μιλήσαμε για τις ε, εκδηλώσεις αυτές για τα 30 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνομπίλ. Αυτή τη φορά στο Όστρεβιτς τι κάνουμε, ξυπνάμε φαντάσματα. Μην ξεχνάμε και την Φουκουσίμα. Τα πυρηνικά ατυχήματα Σκοτών τους πάντες, δεν σέβονται σύνορα. Σκοτώνουν άνδρες και γυναίκες παντού ανά τον κόσμο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας παντού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το θέμα των πυρηνικών αντιδραστήρων και στο έδαφος της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί για να πληρούνται οι συνθήκες της Euratom θα πρέπει να εξυγχρονιστούν πολλοί πυρηνικοί σταθμοί και να δαπανηθούν πολλά δις. Δυστυχώς η Επιτροπή νύπτει τα υπέβαλα ερωτήσεις προς τον κύριο ε, Αρίας Κανιέτε σε σχέση με τον πυρηνικό σταθμό του Αλμαράσα. Η Επιτροπή μου είπε ότι θα το κοιτάξει και θα αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια της νέας οδηγίας. Όμως οι Ισπανικές αρχές μας αναφέρουν ότι όλα λειτουργούν καλώς. Και τη στιγμή που έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε αυτό το σταθμό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να πιστέψω ότι η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για την ασφάλεια και του Αλμαράς και όλων των πυρηνικών σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φένκελ. Κύριε Επίτροπε, μιλάμε για πυρηνικά εργοστάσια τα οποία υποτίθεται ότι δεν είναι ασφαλή. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω κάποια πιο ασφαλή υποτίθεται. Η γερμανική κυβέρνηση δρώντας πανικόβλητη αποφάσισε να κλείσει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια. Ε, υπέπεσε όμως σε αντιφάσεις. Ε, εμφανίζεται λοιπόν η κυρία Μέρκελ ως ε, διασώστης του κλίματος αλλά δεν χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία. Η η αρχή αρμόδια στη Γενέβη λέει πως τα γερμανικά εργοστάσια είναι από τα ασφαλέστερα στον κόσμο, αλλά ειδικά αυτά κλείνουν. Πρώτα απ' όλα ήθελε να είναι η γερμανική κυβέρνηση ε, να είναι πρώτο πόρος, τώρα δεν κάνει τίποτα. Η Γαλλία θα παρατείνει την διάρκεια ζωής των εργοστασίων της κατά 10 χρόνια, θα χτίσει καινούρια. Φιλανδία, είπα, Μεγάλη Βρετανία επίσης θα χτίσουν καινούργια. Στο Βέλγιο ήδη ξανανοίγει ένα πυρηνικό εργοστάσιο που είχε κλείσει μετά τη Φουκουσίμα πάνω στα γερμανικά σύνορα. Η Ιαπωνία ξαναφέρνει σε λειτουργία και στο δίκτυο τα περνικά εργοστάσια που είχε κλείσει μετά την Φουκουσίμα. Η Κίνα χτίζει επίσης. Μέχρι και το Σουδάν θα χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο πάνω από 400 πυρηνικά εργοστάσια από τη Φουκουσίμα και μετά καινούρια. Τι έχουμε στη Γερμανία, μόνο αύξηση των τιμών του ρεύματο. Η πολιτική λοιπόν της Γερμανίας δεν είναι μόνο μη αλληλέγγυα απέναντι στους γειτονέ τη, αλλά οδηγεί και σε ανασφάλεια, σε ψηλότερες τιμές ρεύματος για τους Γερμανούς. α δούμε το παράδειγμα τη Σουηδία και ας πάρουμε πίσω αυτή την απόφαση ε, απόσυρσης από την πυρηνική ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χένκελ, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπούχνερ. Την δέχεστε? Κύριε Μπούχνερ. Κύριε Χένκελ, ήθελα να σας ρωτήσω. Γνωρίζετε πόσο τις εκατό της παγκόσμιας ενέργειας παράγεται σήμερα, κατα, καλύπτεται σήμερα από πυρηνική ενέργεια. Μπορείτε να πείτε όντω ότι συνεισφέρει στην προστασία του κλίματος είναι λιγότερο από 3%. Δεύτερη ερώτηση. Επειδή λέτε ότι είναι τόσο σίγουρα τα γερμανικά εργοστάσια, τι έχετε να πείτε για τις περιπτώσεις Κρούμελ και Μπρουντσπίτελ. Ναι, σας είπα ήδη πως ο αριθμός των πυρηνικών εργοστασίων στον κόσμο αυξάνεται. Στην Κίνα φτιάχνουν 25 καινούρια νέα εργοστάσια. Είναι απλό. Ε, νομίζω είναι σαφές σε όλους ότι δεν εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα, έτσι. Και αυτά τα οποία αναφέρατε τα περιστατικά δεν έχουν σχέση με τον αντιδραστήρα και τα στοιχεία το δείχνουν. Είναι μακράν τα ασφαλέστερα του κόσμου τα γερμανικά πυρηνικά εργοστάσια. Σας ευχαριστώ κύριο Σελίμοβιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Λευκορωσία κατασκευάζει το δικό της αντιδραστήρα με τη βοήθεια της Ρωσίας. Η Ρωσία θα κατασκευάσει όλη την εγκατάσταση. Και 1,5 δισεκατομμύρια κορώνες σφυδικές θα δαπανηθούν σε πρώτη φάση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Όλα αυτά μια στιγμή κατά την οποία η Λευκορωσία ήδη εξαρτάται από ένα και μοναδικό προμηθευτή ενέργεια στη Ρωσία η Ρωσία χρησιμοποιεί σαν όπλο επιρροή στην ενέργεια για να επηρεάζει τις άλλες χώρες για να μπουν στην επιρροή του Κρεμλίνου όπως στην Αρμενία, Καζακστάν, Πολωνία, Ουκρανία, Εστονία, Λετωνία, Γεωργία και αύριο θα γίνει το ίδιο και στη Λευκορωσία. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει αυτό το όλο εγχείρημα διότι αυτό έχει τεράστιες συνέπειες και για τις άλλες χώρες. Και επειδή το έργο αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με το στόχο της ποικιλομορφία των πηγών ενεργείας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαφορεί, πρέπει να σταθμίσει τις γεωστατηγικές συνέπειες αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε κυρία Σάντσες. Ευχαριστώ κύριε Βαλκάρθελ. Η τραγωδία του Τσέρνομπιλ έπληξε δύο εκατομμύρια Λευκορώσους όπως ξέρετε, τα πυρηνικά ατυχήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Μας πλήττουν όλους. Δεν ε, αντλήσαμε τα σωστά διδάγματα, διότι η Λευκορωσία δημιουργεί ένα νέο σταθμό χωρίς να λάβει υπόψη τις αποτιμήσεις ε, στο περιβάλλον, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη και τις δοκιμές αντοχής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ενεργειακό μοντέλο έχει αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίμιση των πυρηνικών καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παραδείγματα όπως τη Γερμανία που θα απομακρυνθούν από τα πυρηνικά και γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ας αρχίσουμε με την, με Καρόνια και το Αλμαράθ στην Ισπανία, να καταργήσουμε αυτούς τους σταθμούς, διότι αυτό θα ήταν καλό για τη ζωή μας, αλλά και για ολόκληρη τη γη. Ο κύριος Ζαόρ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε πολλά σημαντικά σημεία σε σχέση με το σχέδιο αυτό πυρηνικής μονάδας στη Λευκορωσία. Παρόλο όμως που ασχολούμαστε με αυτή την κατασκευή κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα θα πρέπει να μας απασχολήσει και μια κατάσταση εντός των σύνορων. Στην Ουγγαρία δύο νέα τέτοια μπλοκ θα θα κατασκευαστούν τα επόμενα δύο χρόνια από τη Ρωσία όπως ισχύει και με τη Ρωσία, δηλαδή αντιδραστήρες τύπου, ρωσικού τύπου. Αυτοί οι αντιδραστήρες δεν ερμηνεύουν πάρα πολύ ευέλικτα το, κοινωνικό, το πλαίσιο. Σε σχέση με αυτό τον αντιδραστήρα στην Ουγγαρία ασκήθηκε βέτο από τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχει παραβίαση και στα πλαίσια του διαγωνισμού με βάση τις δημόσιες προμήθειες. Διενεργούνται έρευνες για τον τρόπο ανάθεσης. Γιατί ίσως υπήρξε και κρατική ενίσχυση και επίσης υπήρξε και ένα πιλωτικό σχέδιο χωρίς διαφάνεια. Όμως αυτό το κράτος μέλος δεν έλαβε υπόψη τα πυρηνικά απόβλητα, το νόμο δηλαδή περί πυρηνικών απόβλητων. Θα δεχόσαστε να αγοράσετε το οτιδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους και θα μπορούσατε να δεχτείτε την κατασκευή ενός ε, πυρηνικού, μιας πυρηνικής μονάδας ε, στο κέντρο της Ευρώπης. Κύριε Ζάβορ, έχετε μπλε κάρτα. Κύριε Γιάκοβιτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το 1996, όπως ξέρετε, η Κροατία υπέγραψε τη σύμβαση ΕΣΠΟ. Και αυτό το λέω επειδή Μόλις αναφερθήκατε σε λεπτομέρειες που είναι πολύ γνωστές σε μας για το τι συμβαίνει στην Ουγγαρία και αυτού του νέου πυρηνικού αντιδραστήρα στην καρδιά της Ευρώπης. Νομίζω ότι και η Κροατία θα πρέπει να εμπλακεί στις αποφάσεις αυτές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κοινή πολιτική όταν μιλάμε για πυρηνική ενέργεια, μια μελλοντική στρατηγική δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειαζόμαστε πιο ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Δέκα κράτη-μέλη έχουν ε, υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΟ. Νομίζω όμως ότι δεν προσδίδουν τη δέουσα σημασία τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία και η Αυστρία μίλησαν ε, με μεγάλη ανησυχία για αυτό το σχεδιασμό. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη και την Κροατία να είναι περισσότερο δραστήρια και σε μικρότερες χώρες όπως η Ουγγαρία που δεν είναι μεμονωμένο κράτος μέρος. Και ο Σπιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πυρηνική ενέργεια είναι μεν μια ασφαλή μορφή ενεργεία, όμω για να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για ειρηνικού σκοπού θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά μέτρα ασφαλεία ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται όταν ε, εγκαθίστανται ε, πυρηνικοί σταθμοί ή άλλες εγκαταστάσεις ε, κοντά στα σύνορα με την ευρωπαϊκή ένωση. μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο όστροβετς της λευκορωσίας για τον οποίο υπάρχουν επιφυλάξει σχετικά με το εάν και κατά πόσον έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τι υψηλέ προδιαγραφέ ασφαλεία που εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή ένωση. αυτή η περίπτωση φέρνει επίση την επιφάνεια και την ασφάλεια που πρέπει να πληρούν οι πυρηνικέ εγκαταστάσει που προτίθεται να κατασκευάσουν στι χώρε του η αλβανία τα σκόπια και η τουρκία. ιδιαίτερα η τουρκία είναι μια χώρα επικίνδυνη για πρόκληση πυρηνικού ατυχήματο διότι όπω και η λευκορωσία δεν έχει διαφανεί διαδικασίε Προσωμειώσεω ακραίων καταστάσεων πυρηνική ασφαλεία και από την άλλη πλευρά είναι και χώρα σεισμογενή. γι' αυτό η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί ώστε να εξασφαλίσει πω τόσο ο πυρηνικό αντιδραστήρα όστροβε όσο και αυτοί που θα κατασκευαστούν στι χώρε που προανέφερα θα πρέπει να λειτουργούν με τι προδιαγραφέ ασφαλεία που ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι λυπούμε για το ότι ο κύριος Έθριτς έφυγε από την Ολομέλεια και δεν έδειξε ενδιαφέρον στην σοβαρή αυτή συζήτηση. Ε, δείχνει άγνοια όταν λέει ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στις προδιαγραφές του ΟΗΕ για να είμαστε ασφαλείς. Δεν ξέρει πως η ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η ΕΕ, δεν υποστηρίζει το Διεθνές Δικαστήριο του ΙΕ. Τι θα κάνουμε λοιπόν κύριε Θρίτζη, εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για το ότι επαγρυπνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και η Λευκορωσία οπωσδήποτε πρέπει να κάνει τις αξιολογήσεις εκείνες του περιβαλλοντικού αντικτύπου και τα τεστ εκείνα που απαιτούνται από τις διεθνείς ε, συμφωνίες ε, έτσι ώστε και οι γειτονικέ της ε, χώρες αλλά και παραπέρα να είναι ασφαλείς και περιλαμβάνει αυτό και τη δικιά μου τη χώρα και του κυρίου Έθριτς. Υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα όμως. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και κάποιο κόστος στην πυρηνική ενέργεια που δύσκολα υπολογίζονται. Οι ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικέ καταστροφέ σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματο είναι πραγματικά φρικιαστικέ. και έχω δει από πρώτο χέρι εγώ το πώς σημαδεύτηκαν οι ζωές των επιζώντων της ε, Φουκουσίμας, ε, το πώς... Ε, τι να σας πω δηλαδή, δεν μπορούσαν να βγουν τα παιδιά έξω να παίξουν. Από όταν λοιπόν εξελέγνε εγώ έχω συνεργαστεί με ένα δίκτυο πυρηνικής διαφάνειας το οποίο ζητάει περισσότερη ασφάλεια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πως πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια και να στηρίζουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προσπαθούν να το καταφέρουν. Πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος λαμβάνει τεράστιες επιδοτήσεις από τον δημόσιο τομέα, οπότε οφείλει να συνεργαστεί με τις αρχές και με την δική μας ΜΚΟ για να δούμε αν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ, ε, μην μιλάτε με τέτοια ταχύτητα, αλλά να τηρείτε και το χρόνο σας. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα πυρηνικά ατυχήματα φέρνουν θανάτους, πολλές γενναίες ε, αρρώστων και σταματούν τη ζωή. Αυτό το είδαμε μετά από την καταστροφή του Τσερνομπίλ, ιδιαίτερα μετά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οποιαδήποτε κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα θα πρέπει να υπόκειται αυστηρούς ελέγχους. Σήμερα μιλάμε για τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Όστροβετς που κατασκεύασαν οι Ρώσοι και που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να, μειωθεί η εξάρτηση της Λευκορωσίας από τη Ρωσία. Αυτό προβάλλεται, αλλά είναι εσφαλμένο και ψευδές γιατί ο πυρηνικός αντιδραστήρας έχει κατασκευαστεί από Ρώσους Μιλάμε για 2,2 δις δολάρια, όπου συμμετείχαν μόνο ρωσικές κοινοπραξίες. Δεν έγινε καμία μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον για το κατά πόσο μπορεί να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και όλα τα σχετικά. Εμείς μάθαμε για την κατασκευή αυτού του σταθμού από άλλες πηγές και αυτό δεν είναι σωστό. Μαθαίνουμε τώρα ότι και στην ε, Ουγγαρία συμβαίνει το ίδιο με ρωσική χρηματοδότηση, άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τη δική μας ασφάλεια. Με συγχωρείτε, έπρεπε να σας ε, διακόψω γιατί υπερβήκατε κατά πολύ το χρόνο σας. Ο κύριος Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το θέμα το οποίο συζητάμε δεν είναι τεχνολογικό ζήτημα, πρόκειται για ζήτημα το οποίο βεβαίως έχει λυθεί σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία με την σύμβαση ΕΠΣΟ και εφόσον υπήρξε η απαραίτητη κοινοποίηση της κατασκευής του νέου εργοστασίου η Λευκορωσία ε, έχει εκπληρώσει τις ε, τυπικές της υποχρεώσεις. Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διεθνείς ε, προδιαγραφές, μπορεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Αλλά με βάση την σημερινή δήλωση θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνει παρά τα αιτήματα που υπάρχουν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, Ουκρανία όπου παρατάθηκε η περίοδος λειτουργίας ε, ποινικών δεθείων μέχρι το 2030 παρά το ότι θα έπρεπε να έχουν ήδη κλείσει. Είναι ζήτημα αρχής να έχουμε τις ίδιες αρχές για όλους. Και επίσης δεν έχει ακόμα κυρωθεί το πρωτόκολλο του Κιέβου τόσα χρόνια μετά την υπογραφή του. Μιλάμε για πάνω από 17 αντιδραστήρες και άλλου 4 οι οποίοι σχεδιάζονται. Σα ευχαριστώ κύριο Μπούχνερ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πυρηνικό εργοστάσιο του Οστροβέτς που κατασκευάζεται στην Λευκορωσία παραβιάζει διάφορες διεθνείς συνθήκες. Παραδείγματο χάρη τη σύμβαση του Άρχους, παραδείγματο χάρη ναι, την υποχρέωση να γίνουν stress τεστ. Εσείς θα αγοράζετε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ πως ο τύπος WWR 1200 εγγενώς δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας γιατί η σχέση μήκους προς διάμετρο του ίδιου του αντιδραστήρα είναι προβληματική. Οπότε η Λευκορωσία δεν έχει αυτή την στιγμή τους οικονομικούς πόρους για να κάνει κάτι καλύτερο. Όσον αφορά λοιπόν την ε, ασφάλεια ε, και βεβαίως όσον αφορά και την διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε εσείς κύριε Επίτροπε να μας εγγυηθείτε πως ε, θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει μόνο της Λευκορωσία. Κύριε Σάντζη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 26 Απριλίου είχαμε την 30η επέτειο του Τσερνομπίλ. Και η Λευκορωσία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της υπόθεσης αυτής ε, και βλέπετε πως ε, τα αποτελέσματα διαρκούν ακόμα και σήμερα και έχουμε πραγματικά μια απόδειξη για το ότι μιλάμε για ένα διασυνοριακό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πέρα από τα σύνορά μας και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είναι ασφαλές αυτό το ποινικό εργοστάσιο. Έχει και μια πολιτική σημασία το ζήτημα γιατί η Λευκορωσία εξαρτάται από τη Ρωσία. Η ενεργειακή εξάρτηση και η ενεργειακή ασφάλεια της ε, ε, Λευκορωσίας ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί στον 21ο αιώνα αλλά η Ουγγαρία επιστρέφει στο παρελθόν με την ε, τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται τώρα στον ε, αντιδραστήρα POX 2. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να επιστήσω την προσοχή της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου στο ότι θα πρέπει να ξέρουμε και το τι γίνεται στην Ουγγαρία. Κάθε νέο πυρηνικό εργοστάσιο είναι τελικά άλλο ένα πρόβλημα γιατί υποτίθεται ότι προσπαθούμε να διαδώσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η πυρηνική ενέργεια είναι εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι δεν είναι μια συζήτηση γενικόλογη, είναι πολύ συγκεκριμένη δική συζήτηση. Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να συζητούμε την δομή του εφοδιασμού ενεργείας στην Ευρώπη, σε ποιο βαθμό η πυρηνική ενέργεια είναι χρήσιμη, αναγκαία κλπ. κλπ. Πρόκειται περί συγκεκριμένη επενδύσεως, ε, που είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας τόπος μια περιοχή νευραλγικής σημασίας και για τη Λιθουανία και για την Πολωνία. Και ομολογώ ότι εκπλήσωμε κάπως από την απάντηση του κυρίου Επιτρόπου που μιλάει σαν να μην πρόκειται παρά μόνο μια ακόμα επένδυση που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τεχνικής απόψεως. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην καταστροφή του Τσερνομπίλ. Εμείς ήμασταν την άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος. Ξέρουμε τι σημαίνει έλλειψη σεβασμού για το περιβάλλον. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και βέβαια, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματο είναι κάτι που δημιουργεί πολλές αμφιβολίες. Πολλές φωνές ακούστηκαν που υπογράμμισαν το ρόλο της Ρωσίας. Πρόκειται περί επενδύσεως που συγχρηματοδοτείται από τη Ρωσία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ρωσικές επενδύσεις έχουν σκοπούς πολιτικούς. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να φροντίσει την ασφάλεια όλη τη Υπήρου και να ασκήσει πραγματική εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να αποσιωπεί το γεγονός ότι πρόκειται περί ρωσικής επενδύσεως για πολιτικούς σκοπούς. Πράγματι, στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Θεογιούσκη. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν με ενδιαφέρει από πού έρχονται τα χρήματα για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Λευκορωσία. Δεν με ενδιαφέρει αν η Λευκορωσία μετά θα ξαναπολύσει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτό το σταθμό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα πυρηνικά απόβλητα. Η ασφάλεια της παραγωγής. Θα είμαστε σίγουροι, θα είμαστε ασφαλείς στη ζώνη εκεί γύρω από την περιοχή του εργοστασίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ξεκάθαρα ότι τα θέματα ασφαλείας που αναφέρονται στο ερώτημα που υπευλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξηγηθούν, πραγματικά να εξηγηθούν. Όσον αφορά τι οικονομικέ πτυχέ, αυτέ είναι διαφορετικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στη διάθεσή της για να ερευνήσει και να ελέγξει αυτό το κατασκεύασμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Λευκορωσία είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της πρώην Έσου και ο διπλωματικός προσανατολισμός της κυβέρνησης Λουκατσένκο προς τη Μόσχα δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο για δημιουργία αρνητικού κλίματος με οποιαδήποτε αφορμή. Προφανώς και ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος δεν περιορίζεται στα σύνορα των κρατών το γνωρίζουμε πολύ καλά από το ατύχημα του τσερνόμπιλ και προφανώς η κυβέρνηση της λευκορωσίας καθώς και όλοι οι ηθήνοντες που εμπλέκονται στην κατασκευή του νέου πυρηνικού εργοστασίου στο αστραβέτς πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μονάδα να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της διεθνούς οργάνωσης πυρηνικής ενέργειας. το ίδιο όμως πρέπει να συμβεί και για την τουρκία που επιχειρεί αντίστοιχα να οικοδομήσει πυρηνικό εργοστάσιο απέναντι από τα δωδεκάνησα σε μια άκρος σεισμογενή περιοχή επίσης υπάρχουν μια σειρά από παλιά εργοστάσια στη δυτική ευρώπη των οποίων η λειτουργία πρέπει να μας ανησυχεί. πότε θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό συνολικά; πότε θα συζητήσουμε για τις μονάδες της ντοέλ και του τιάντζ που έπρεπε από το 2015 να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στο βέλγιο; Ευχαριστώ. Η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι ύψης της σημασίας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι το ίμιση των κρατών μελών έχει πυρηνικούς αντιδραστήρες και υπάρχουν κίνδυνοι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε. Αυτό συμβαίνει με το αλμαρά της Ισπανίας που βρίσκεται στο, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Θα πρέπει λοιπόν να κηρυχθεί η πάυση λειτουργίας πολλών πυρηνικών σταθμών για την ανθρώπινη υγεία και να υπάρχει εποπτεία μετά από το κλείσιμό τους. Να δούμε δηλαδή πώς αποθηκεύονται τα ραδιενεργά υλικά πώς ε, μπαίνουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν, όπως και η βιωσιμότητα και η επιπτώση στο περιβάλλον. Ρότ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βέβαια, η κατάσταση στη Λευκορωσία σχετικά με την πυρηνική ενέργεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε και σε επίπεδο διεθνές. Και είναι σημαντική επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Από την αρχική μας συζήτηση είδα ότι υπάρχει και θέμα αρχής που προβάλαμε στη συζήτηση. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί διεθνείς οργανισμοί και φορείς πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους υποστηρίζουμε τους φορείς. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη Διεθνή Οργάνωση Πυρηνικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, που παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Και σε ευρύτερο πλαίσιο ε, για άλλες πολιτικές. Στους G7, του G20, το ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό τη Διεθνή Οργάνωση για Τυποποίηση, το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο ΑΣΕ, Ιντερπολ και του άλλου φορεί έχουμε. Είναι οργανισμοί που θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται να εστιάζεται συζήτηση επί ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και λένε ότι αν φύγουμε θα είμαστε απομονωμένοι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε. Ο κ. Συναδεινός. Η κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Όστροβετ τη Λευκορωσία έχει τεράστια σημασία για την ενεργειακή πολιτική τη Λευκορωσία αλλά και τη Ένωση, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και προστασία του πυρηνικού σταθμού και του περιβάλλοντο. Είναι προφανέ ότι η λευκορωσία έχει κάθε δικαίωμα να αναζητήσει εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια αν αναλογιστούμε ότι το 90% του αερίου που χρησιμοποιεί εισάγεται από τη Ρωσία. Βέβαια, οι φωνέ διαμαρτυρία που ακούγονται αφορούν στη συμφωνία τη Λευκορωσία με τη ρωσική εταιρεία για την κατασκευή του σταθμού και τη μελλοντική διαχείριση αποβλήτων, αλλά και στη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματο με 22 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία. Νομίζω ότι η Λευκορωσία ω κυρίαρχο κράτο μπορεί να υπογράφει ενεργειακέ συμφωνίε χωρί υποδείξει και απαγορεύσει περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί η διενέργεια προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων η πληρότητα των προτύπων ασφαλεία και η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά του παρακείμενου ποταμού νέρη. σε αυτό μπορούμε να συνδράμουμε τις αρχές της λευκορωσίας, αλλά και τη διεθνή υπηρεσία ατομική ενέργεια με την ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών φορέων πυρηνική ασφάλεια. ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλό διακύβευμα όταν μιλάμε για ασφάλεια στο, στη χρήση των πυρηνικών. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα από τα ευρύτερα ζητήματα που εφήγησαν. Στην περίπτωση του Στράβετς θα ήθελα να σας πω αυτό που είπα εξ αρχής η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς και να τηρούνται φυσικά. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Γι' αυτό η προτεραιότητά μας τώρα είναι να ε, τεθεί έγκαιρα σε εφαρμογή η κατάσταση δοκιμών, στο, οι στον σταθμό Όστροβετς. Η Επιτροπή θα σας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για οποιασδήποτε εξελίξεις. Ορισμένες ή πολλές από τις λύσεις στο ζήτημα αυτό σχετικά ταυτίζονται με το τέλος του πυρηνικού απομονωτισμού και απομόνωσης ως προς την ε, ενεργειακή αγορά και τη δική μας, της Λιθουανίας αλλά και όλων των βαλτικών κρατών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως στην ενεργειακή οικονομία της Ευρώπης. Τα καλά νέα είναι ότι επιτελείται πρόοδος Πρόσφατα αρχίσαμε τις ε, διαδικασίες για την ε, ηλεκτρική συνδεσιμότητα της Λιθουανίας με την Πολωνία και την Σουηδία μέσω του Μπαλτ έτσι ώστε να υπάρξει διασυνδεσιμότητα με ολόκληρο το ηλεκτρικό ε, δίκτυο. Ιδιαίτερα στις βαλτικές χώρες που αυξήθηκε από 4% σε 22%. Στο φυσικό αέριο Γίνεται, γίνονται έργα για τη διασυνδεσιμότητα ε, Πολωνίας-Λιθουαμίνιας. Ε, GIPL ονομάζεται και είναι ο, η πρώτη, ο πρώτος σύνδεσμος ε, φυσικού αερίου μεταξύ Ανατολικής Βαλτικής και Ευρώπης και όταν ολοκληρωθεί το 2019 δεν θα υπάρχει απομόνωση ως προς τη χρήση του φυσικού αερίου σε αυτή την περιοχή. Θα έχουμε και νέους ε, διάβλους φυσικού αερίου έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της πρόοδου αφορά το σχέδιο συνδεσιμότητας ε, των βαλτικών χωρών στον τομέα του φυσικού αερίου έτσι ώστε να συνεργαστούν όλες οι χώρες και να ενταχθούν αυτές οι περιφέρειες στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους για το τι μπορούμε να επιτύχουμε βάσει την ε, Ένωση στον τομέα της ενέργειας. Η επόμενη πρόκληση είναι να υπάρξει συγχρονισμός δράσης βαλτικών κρατών και άλλων απομονωμένων περιοχών με την ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύουμε στην Ενεργειακή Ένωση που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη, όπου θα μιλάμε με μία φωνή προς τους εξωτερικούς εταίρους μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των αναγκών των Ευρωπαίων. Γι' αυτό η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι θα συμβαδίσουμε στην προσπάθειά μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε όλα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικότητα, να υλοποιηθούν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Λίγη λοιπόν η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή έχουμε σύντομες παρουσιάσεις εκθέσεων και η πρώτη είναι της κυρίας Χόιμπουχ για τη νέα συμμαχία για την επιστηστική ασφάλεια και τη διατροφή. Η εισηγήτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.